μέρες αυτής της διαδικασίας θα δημοσιευθούν στα πρωτόκολλα αυτής της ε, συνεδρίασης. Ο κύριος Χέλμουτ Σόλτ θα αντικαταστήσει τον Μίκαλ Γκούσταυσον με ανακοίνωσή της η μας ενημερώνει για αυτήν την αντικατάσταση. Υπάρχει κάποια αντίρρηση όσον αφορά αυτή την αντικατάσταση. Όχι, λοιπόν, θεωρούμε ότι ο κύριος Σόλτς παίρνει τη θέση του κύριου Γκούσταυσον.